Τώρα συνεχίζουμε με την έκθεση του κυρίου Γκίγκολτ για Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ιδιαίτερα του Σκιώδη, τον κύριο Σάντσεθ Πρεσέδο και την κυρία Λούλινγκ. Ε, να σας ευχαριστήσω θερμά για την καλή συνεργασία που είχαμε για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης γιατί ήδη πριν από τρία χρόνια σε ένα κάπως διαφορετικό πλαίσιο είχαμε ασχοληθεί εντατικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκών εποπτικών οργάνων για τη χρηματοπιστωτική εποπτεία ε, και τότε έγιναν 26 τρίλογοι με το Συμβούλιο και υπήρξαν μακρές διαδικασίες για το πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε και να κάνουμε αποτελεσματική την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή ώστε να μπορέσει να οδηγεί σε μια αποτελεσματική εποπτεία. Και μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις ε, καταλήξαμε μετά από τρία χρόνια, κάναμε ένα απολογισμό και έχουν εκπονηθεί μελέτες καταρχήν για τις ε, τομεακές ε, αρχές εποπτείας για ασφάλειες, αγορές και τράπεζες και από την άλλη τη μακροπροληπτική εποπτεία. Και το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον και ήταν πολύ κοντά σε αυτό που είχαν ε, βρει οι παραπλήσιες έρευνες ευθύνες της ε, Κομισιόν. Πραγματικά οι υποπτικές αρχές ε, δούλεψαν σωστά, εκπλήρωσαν την εντολή τους, ιδιαίτερα όσον αφορά την νομοθεσία, αλλά όταν πρόκειται για άλλα δικαιώματα τα οποία τους ε, εκχωρήσαμε, οι υποπτικές αρχές πολύ συχνά δεν μπόρεσαν να κάνουν τη δουλειά τους. Για παράδειγμα, όσον αφορά τη μη εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου σε πάρα πολλές χώρες, μέλη, όπου τελικά δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί. Και το ίδιο ισχύει για την δεσμευτική διευθέτηση, τη θυσία των διαφορών. Ε, ε, εδώ η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή δεν ε, χρησιμοποιείται για την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών. Με άλλα λόγια, οι, έρευνα, οι έρευνες μάλλον διαπιστώνουν ότι δεν προχωρήσαμε τόσο πολύ όσο επιθυμούσαμε ε, κατ' ουσία. Και η μακροπροληπτική εποπτεία, η οποία είναι σημαντική όσον αφορά την επισήμανση συστημικών κινδύνων, εδώ διαπιστώσαμε ε, πολλές αδυναμίες. Για παράδειγμα, είναι πολύ μικρότερη αρχή από ότι η αντίστοιχη αρχή των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει στο επίπεδο της πρόληψης, ίσως επειδή βρισκόμαστε ε, στο επίκεντρο της κρίσης. Αλλά πέρα από αυτή τη διάγνωση, η έκθεση λέει ξεκάθαρα ε, ότι μπορούν να γίνουν κάποιες συστάσεις. Ε, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση, ανεξάρτητα από τις εθνικές εποπτικές αρχές, να λαμβάνει αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή ε, χωρίς ε, μία απόφαση στο Εποπτικό Συμβούλιο των Εθνικών Εποπτών δεν είναι δυνατόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ξεκινήσουν να κανουν μια διαδικασία εργασίας. Ε, και εδώ θέλουμε να είναι οι εθνικές αρχές να είναι πιο ανεξάρτητες ουτε ώστε οι εθνικοί επικεφαλείς να μπορούν να ξεκινήσουν μια διαδικασία νομικής παραβίασης σε εθνικό επίπεδο. Εν γέννη η έκθεση περιλαμβάνει πολλές προτάσεις εν σχέση με το πώς θα μπορούμε να ενισχύσουμε την εξουσία τη Ευρωπαϊκή Εποπτική αρχή. Και επιπλέον ε, προτείνουμε οι προσβάσιμε πληροφορίε να απλουστευτούν και όλε οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές θα πρέπει να έχουν δεδομένα όπω και οι εθνικέ εποπτικές αρχέ και θα πρέπει να υπάρξει μια εναρμόνιση ούτω ώστε οι οικονομικέ επιχειρήσει να μην αντιμετωπίζουν πολύ με υψηλό κόστο. Και εν γέννη θέλουμε μια ενίσχυση της ε, ε, χρηματοδότησης των υπηρεσιών αυτών. Ε, η Κομισιόν έχει ένα χρόνο να ακολουθήσει αυτές τις συστάσεις ή να αιτιολογήσει γιατί δεν το πράττει. Ε, αναμένουμε λοιπόν ε, τις αποφάσεις της Επιτροπής και πραγματικά θα μας χαροποιούσε ιδιαίτερα αν ε, πολλές από τις προτάσεις μας τις οποίες επεξεργασήκαμε σε μεγάλο βαθμό ομόφωνα τελικά μπορούν να υιοθετηθούν στο δικό σας κείμενο κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε ο λόγος στην κυρία Λούλιν. Πρέπει να πω, όπως και συγητής, εγώ δεν βλέπω μόνο τις τρύπες στο τυρί, για να το πω έτσι, σε ό,τι αφορά τη δουλειά και τις επιδόσεις των ευρωπαϊκών αρχών, αλλά κατά την πρώτη ανταλλαγή απόψεών μας για την έκθεση πρωτοβουλία αυτήν, πριν από 7 μήνες, είχα θέσει ένα αμφιβόλο την όλη χρησιμότητα, το σκόπιμον αυτής της διαδικασίας, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όφιλε τον Γενάρη κιόλα του 2014 να υποβάλει τη δική της έκθεση για τη λειτουργία των τριών αρχών εποπτείας που δημιουργήθηκαν το 2010. Επιπλέον πρέπει να γνωρίζουμε και να μην ξεχνούμε ότι η Ευρωπαϊκή Εποπτεία ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πλήρη αναδιάρθρωση με την ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Τραπεζική Ένωση που αυτή τη στιγμή οικοδομείται. Δεν νομίζω ότι το ε, Ευρωκοινοβούλιο ως ε, συνομοθέτης θα πρέπει να παράγει ένα κείμενο που μοιάζει σαν μια πολλωστή έκθεση οικονομικών συμβούλων διότι εδώ η ουσία βρίσκεται στις λεπτομέρειες. 25 ε, σημεία, 19 αιτιολογικές σκέψεις, 180 εδάφια και ε, πολλαπλέ ερωτήσει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έκθεση αυτή καταντά δυσνόητη. Αδύνατο να την διαβάσει κανεί. Επί του ουσία, λοιπόν πρόεδρε δεν υπήρξε συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων και εγώ πρέπει να πω ότι παραμένω χωρίς ικανοποίηση για την μορφή αλλά και για τα συμφέροντα του Κοινοβουλίου που δεν ε, γίνονται σεβαστά. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σάντσες Πρεζέντο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η δημιουργία Ευρωπαϊκού Συστήματος Εποπτείας το 2010 έγινε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Μεταρρύθμισης και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Γκίγκολτ ε, και τους υπόλοιπους εισηγητές γιατί ε, στηρίζεται στην πρώτη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την ε, ΕΑΚ. Ε, προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια, η ανεξαρτησία και η αποτελεσματικότητα του συστήματος μέσω άμεσης πρόσβασης και ανταλλαγής πληροφοριών χωρίς επικαλύψεις, ενίσχυση του ρόλου του Προέδρου, και βελτίωση της συνεργασίας των ενεχόμενων μερών. Ε, το να ενισχυθεί η εντολή ε, για την ενίσχυση των θεσμικών οργάνων με βρίσκει σύμφωνο. Επίσης να ενισχυθεί η δυνατότητα ειρηνικής διαθέτησης των διαφορών. Θα πρέπει, ε, με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και θα εδραιωθεί η ισότητα μεταξύ των χωρών μελών μέσω της θέσπισης ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού ε, και ε, μπορεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή. Ah, yes. Do you want Θέλετε να δεχτείτε μια ερώτηση από τον κύριο Ντόρκμουντ. Εντάξει. Κύριε πρέσέδα Πρεσέδα, ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε την ερώτησή μου. Αναφέρατε ότι η μετάφραση αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και διαφάνεια ότι αυτό αναφέρθηκε από τη μετάφραση αλλά κατ' εσάς Αυτές οι έννοιες συμπεριλαμβάνουν και το ρόλο του Λιξεμβούργου ως ε, φορολογικού παραδείσου ή όχι. Ναι. όχι. Όχι, δεν τελείωσα. Είναι επομένως θεμητό ο κύριος Σαντέρ να θεωρείται ως ε, υποψήφιος πρόεδρος της Κομισιόν όταν έχει το σε αυτές τις δραστηριότητες φοροαποδιαφυγής ως φορολογικός παράδεισος. Νομίζω ότι είναι τα πολιτικά κόμματα και οι πολίτες αυτοί που θα πρέπει να θεσπίσουν τις δημοκρατικές διαδικασίες και εγώ βεβαίω είμαι υπέρ του ότι οι αρχές αυτές ε, που να λειτουργούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής και βεβαίω να ανταλλάσσουν αυτόματα τα δεδομένα γιατί με τον τρόπο αυτό μπορεί να μειωθεί το κόστος και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των πλευρών. Ο κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για πολύ σημαντικό θέμα και πρέπει να συγχαρούμε τον κύριο Γκίγκουλτ καθώς και την κυρία Λούλινγκ η οποία είναι τώρα 85 ετών και είναι η τελευταία σύνοδος στην οποία συμμετέχει. Ευτυχώ αυτή τη στιγμή η Ιρλανδία ανακάμπτει μετά από τη μεγάλη κρίση, αλλά αυτό που έφταιγε δεν ήταν η έλλειψη νομοθεσίας, αλλά η κακή εφαρμογή της. Και αυτό οφειλόταν με τη σειρά του στην κακή εποπτεία. Άρα χρειάζονται πανενωσιακοί κανόνες εποπτείας. Πρώτον, για να πάρουμε τα μαθήματα από αυτά που έχουν γίνει και δεύτερον, για να φανεί ότι οποιοδήποτε και να χειρίζεται τα θέματα πάντα χρειάζεται και κάποιος πάνω από εκείνον για να εποπτεύει. Έτσι θα υπάρξει εγγύηση συνέπειας και ο, του ότι όλοι θα κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει. Ευχαριστούμε πολύ. Λίγη αυτή η συζήτηση. Πρέπει όμως τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Πόρκ, τον Επίτροπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Γκίγκολτ, την Επιτροπή σα και το Ευρωκοινοβούλιο συνολικά για τη δουλειά σα στην έκθεση αυτή για το Ευρωπαϊκό Σύστημα τη Χρηματοπιστωτική Εποπτεία. Η έκθεση τονίζει τη σημαντική συμβολή που έκανε το σύστημα αυτό στην ε, ενίσχυση της ε, εποπτείας στην εσωτερική αγορά. Το ευρωπαϊκό σύστημα της χρηματοπιστωτικής εποπτείας έχει δημιουργηθεί για να αντιμετωπίσει τις ανεπάρκειες, τις ανισότητες και τον κατακαιρματισμό που ίσχυε στην εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην αγορά, όπως αποκαλύφθηκαν μέσα από την κρίση και την έλλειψη συντονισμού μεταξύ εποπτών. Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι μπορέσαμε δεν μπόρεσαν μάλλον οι εποπτές να καλύψουν τις προσδοκίες που τους ε, αφορούσαν. Υπήρξαν βεβαίως τομείς όπου θεωρήθηκε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, όπως η διακυβέρνηση των αρχών, όπου θα πρέπει να επικεντρώνονται περισσότερο στι μελλοντικέ ανάγκε. Ε, εκτιμούμε τη συμβολή της έκθεσης αυτής, γιατί βάσει και τη δική μα αποτίμηση και των διαβουλεύσεων που διεξήγαμε, ε, είδαμε ότι ακρογωνιαίος λήθος είναι η μεταρρύθμιση μετά από τα όσα συνέβησαν με το ξέσπασμα της κρίσης. Χρειάζεται ακριβώς οι αρχές αυτές εποπτείας να συνεχίσουν το έργο τους γιατί έχουν εκπληρώσει τώρα τις υποχρεώσεις τους και έχουν καταφέρει να εξηγιάνουν ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων που είχαμε. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχυθούν περαιτέρω. Εδώ βλέπουμε η έκθεση να μιλά για κάποιε λεπτομέρειε τη λειτουργία ε, του συστήματο χρηματοδοτική εποπτεία. Όμω ε, δεν αμφισβητείται η ανάγκη ύπαρξή του, <coughs> του συστήματο αυτού. Θα συνεχίσει να διδραματίζει σοβαρό ρόλο στην υλοποίηση τη ευρωπαϊκή νομοθεσία σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά, την εσωτερική αγορά. Πρόσφατα, πρόσφατη θεώρηση για την διακυβέρνηση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι κάτι που συνάδει με αυτό το συμπέρασμα θα πρέπει έτσι κι αλλιώ ε, αυτό το σύστημα να παραμείνει στο κέντρο τη ευρωπαϊκή εποπτεία με ένα διαφορετικό πεδίο και μια σειρά από να καλύπτονται. Η αποξολόγηση των δράσεων αυτών για το σύστημα χρηματοδοτική εποπτεία όπω δημιουργείται η Τραπεζική Ένωση είναι κάτι που θα το χρειαστούμε και θα παρακολουθείτε στενά και στο μέλλον. Εκτιμούμε την συμπολίτη έκθεση αυτή σε κάποια βασικά ζητήματα ω προ τη λειτουργία των αρχών. Λόγω χάρη, συμφωνούμε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να διασφαλίσουμε περαιτέρω ότι όπου λαμβάνονται αποφάσει πρέπει να είναι προ το ευρωπαϊκό συμφέρον. Επίση, συμφωνούμε ότι περαιτέρω εξετασή πρέπει να γίνει ε, των διαδικασιών ευθυγράμμιση, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι οι υποπτικέ αρχέ μπορούν να φέρουν ει πέρα στι αρμοδιότητέ του, λαμβάνοντα υπόψη ε, ε, του δημοσιονομικού περιορισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, συμφωνούμε ότι η διαδικασία λήψη αποφάσεων ε, στο επίπεδο του Γενικού Συμβουλίου του Συστήματο Χρηματοπιστωτική Αποκτήας θα μπορούσε να εξορθολογιστεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, ε, λαμβάνει υπόψη τι ε, επιταγέ της... τα αιτήματα τη έκθεση αυτή και θα φροντίσει να τα υλοποιήσει στον τομέα αυτό. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπόρτ. Η έκθεση, η συζήτηση κλείνει. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στι 12. Επόμενο σημείο η έκθεση της κυρίας Σίντβελτ, πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα και να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για τέσσερα λεπτά. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα της διαφανίας και αρχίζω